Θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Αγαπητέ κυρίε και κύριοι, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, σα ευχαριστώ εξ ονόματο τη Επιτροπή για την ευκαιρία που μα δίνετε σήμερα να μιλήσουμε σήμερα ε, με την ευκαιρία τη Διεθνού ημέρα Ρωμά που εορτάστηκε την περασμένη Παρασκευή. Αυτή οι διακρίσει κατά τον Ρωμά είναι πολύ εξαπλωμένε σε ολόκληρη την Ένωση και είναι μια ε, μορφή ρατσισμού που συνδέεται στενά με αρνητική στερεότυπα και στιγματισμό των Ρωμά και μάλιστα αυξάνεται. Συνδέεται με την αύξηση του ριζοσπαστισμού και των ακραίων τάσεων γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η κατάσταση προκαλεί ανησυχίες. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε στεναρή στάση και να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να πάψουν αυτά τα αρνητικά φαινόμενα που είναι ασύμβατα με τις απόψεις τις οποίες ε, στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει ένα ε, συμπαγές σε πλαίσιο πολιτικών, νομικών και οικονομικών μέσων που αν εφαρμοστούν σωστά θα πρέπει να οδηγήσουν σε αποτελέσματα επιτόπου. Η Κομισιόν έχει επιτείνει τις προσπάθειές της ώστε να εξασφαλίσει τη σωστή εφαρμογή των νομοθεσία κατά του ρατσισμού σε σχέση με τους Ρωμά. Επίσης, καλεί τα κράτη-μέλη να επιδείξουν μεγαλύτερη πολιτική βούληση και οραματικότητα για να καταπολεμήσουν τον ρατσισμό και να ευνοήσουν την ένταξη των Ρωμά. Η ένταξή τους στις πολιτικές παιδείας, αγοράς εργασίας και πολιτικής ζωή είναι, είναι βασικά συστατικό για μια λειτουργική και υγιή κοινωνία. Φέτος έχουμε ξεκινήσει μια στοχευμένη εκστρατεία ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις κατά των Ρωμά. Ονομάζεται για τους Ρωμά με τους Ρωμά συμπεριλαμβάνει κατάρτιση σε στενή συνεργασία με τους Δήμους σε επιλεγμένα κρατημέλη. Η καταπολέμηση του ρατσισμού ε, κατά των Ρωμά και των ε, γύφτων ε, περιλαμβάνεται μέσα στην ετήσια έκθεση της Κομισιόν για την πρόοδο που σημειώνεται για την προώθηση της ένταξης των Ρωμά καθώς και στις συστάσεις του Συμβουλίου για την αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρωμά πρόκειται για τα πρώτα νομικά μέσα της Ένωσης που ρητά αναφέρονται στους Ρωμά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει και υποστηρίζει ε, στεναρά την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ορισμό στις της Δευτέρας Αυγούστου ως ε, ε, ημέρα επέτειο του ε, ολοκαυτώματος των Ρωμά στην Ευρώπη. Είναι καθήκον μας να αναγνωρίσουμε και να θυμόμαστε όλους εκείνους που υπέφεραν υπό το ναζιστικό καθεστώς συμπεριλαμβανομένων των Ρωμά. Οι Ρωμά στα στρατόπεδα συγκέντρωσης αποτελούν ένα φρικτό κεφάλαιο της ανθρώπινης ιστορίας που είναι λιγότερο γνωστό. Η Κομισιόν στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε το ψήφισμα αυτό να έρθει στο Συμβούλιο για περαιτέρω συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ε, Θα δώσω τώρα το λόγο στους ε, συναδέλφους που έχουν ζητήσει να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Θα ήθελα να προβώ σε μία διευκρίνηση. μετά από την έναρξη συζήτηση από πλευρά του Προέδρου. Εδώ δεν γίνονται, σε αυτή τη συζήτηση δεν, προβλέπονται, ε, δεν προβλέπεται συζήτηση κατόπιν αιτήματο, δεν δεχόμαστε μπλε κάρτε, δεν θα υπάρξει κατσδιάη. Σε αυτήν εδώ τη συζήτηση, μόνο οι εγγραμμένοι δηλαδή θα μιλήσουν. Και τώρα θα μιλήσει ο κύριος Όλβενη για τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μεγάλη για μένα που μπορώ να πάρω το λόγο σήμερα σε αυτή την παγκόσμια ημέρα Ρωμά εξ ονόματος του ΕΛΚ. Πρόκειται για ένα θέμα που φυσικά έχει μια κοινωνική, μια ανθρώπινη πτυχή. Μια ιστορική επίσης πτυχή. Το 2011 κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της χώρας μου ξεκινήσαμε μια στρατηγική με επίκεντρο τους Ρωμά. Πρόκειται για την κοινότητα αυτών των ανθρώπων των οποίων θα πρέπει να εξετάσουμε εκ νέου την κατάσταση και να στηρίξουμε την ενσωμάτωσή τους αντιμετωπίζουν επιπλέον δυσκολίες οι Ρωμά εάν θέλουν να ξεπεράσουν τον αποκλεισμό τους, εάν θέλουν να μπορέσουν να ενσωματωθούν στις κοινωνίες μας παρόλο που έχουν διαφορετικές συνήθειες, αντιμετωπίζουν διακρίσεις και προκαταλήψεις από τις κοινωνίες μας. Χρειάζονται λοιπόν οι Ρωμά ειδικέ ενισχύσεις, βοήθεια, αντιμετώπιση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αλλάξει η στάση μας, θα πρέπει να δείξουμε περισσότερο σεβασμό και εκείνη περισσότερη προσαρμοστικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε περίπτωση πρέπει να δημιουργήσει επαγγελματικά πλαίσια έτσι ώστε να στοχεύσει καλύτερα τα ειδικά προβλήματα, τις δυσκολίες και τις ανάγκες αυτής της κοινότητας. Η στρατηγική για τους Ρωμά λοιπόν φυσικά και έχει σαν σκοπό να πάψει να υπάρχει κάθε είδους αποκλισμός, αντιμετώπιση με προκαταλήψεις, ξενοφοβία και ρατσισμό. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν δράσουμε από κοινού μαζί τους με την κοινότητα αυτή και υιοθετήσουμε κοινέ αποφάσεις αν θέλουμε να είναι βιώσιμο αυτό το σχέδιο θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους ίδιους τους Ρωμά. Να λάβουμε υπόψη μας την ιστορία τους, τον πολιτισμό τους που να ενσωματωθεί στα εκπαιδευτικά προγράμματα των χωρών μας, να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους, έτσι ώστε να ενσωματωθούν πραγματικά τα εκατομμύρια των Ρωμά πολιτών της Ευρώπης θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ώστε να δημιουργηθούν ίσες ευκαιρίες από την παιδική ηλικία, από την προσχολική ηλικία, ακόμα και αν οι προσπάθειες αυτές που πρέπει να ξεκινήσουν πολύ νωρίς θα έχουν αποτελέσματα πολύ αργότερα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δώσουμε στα παιδιά των Ρωμά τη δυνατότητα από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους να ενσωματωθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα των χωρών που ζουν. Να ανοίξουμε τις πόρτες των σχολείων μας. Να δείξουμε πνεύμα αλληλεγγύης προς τις κοινότητες των Ρωμά. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για την ε, ευφυΐα της κοινότητας των Ρωμά, να τους επιτρέψουμε να επιτύχουν την ενσωμάτωσή τους, να εργαστούν στις ευρωπαϊκές χώρες που ζουν. Το δίκτυο των κολεγίων Ρωμά είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ενσωμάτωσης παιδιών της κοινότητας Ρωμά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ξεκινήσαμε λοιπόν από κοινού με την κοινότητα των Ρωμά αυτές τις προσπάθειες. Ας συνεχίσουμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Πόστ. Για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πέρσι συζητήσαμε ένα ψήφισμα για την ανάγκη να αναγνωρίσουμε τον ε, ρατσισμό κατά των ε, τσιγάνων και την αναγνώριση του ολοκαυτώματος των Τσιγκάνων στο Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο. Ενεκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία αυτό το ψήφισμα και το Κοινοβούλιο έχει δείξει σαφώ με ποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπίσουμε την απορριπτική στάση σε σχέση με του Ρωμά. Οι Ρωμά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ω ανθρώπινα όντα. Η αντιμετώπιση, η αντική αντιμετώπιση των τσιγκάνων είναι κάτι το οποίο είναι μια, ένα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνεί και η Κομισιόν και το Συμβούλιο και όλοι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό. Αλλά το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτό στην πράξη. Δεν αρκεί να έχουμε κοινωνικά μέτρα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μορφή ρατσισμού που είναι κάτι το πολύ απτό και συγκεκριμένο. Πρέπει να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε αυτή την ε, ιδέα και στο κύριο κορμό της κοινωνίας μας και το κοινοβούλιο μας θέλει να συζητήσει για τα θέματα αυτά, γιατί θέλει να θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα. Τι συγκεκριμένα μέτρα μπορούν να πάρουν τα κρατη για να αντιμετωπίσουν αυτή τη συγκεκριμένη μορφή ρατσισμού κατά τον Ρωμά. Το Συμβούλιο και τα κρατη θα πρέπει να θέσουν συγκεκριμένου και φιλόδοξου στόχου για το έργο του, ώστε η Κομισιόν <clears throat> να μπορέσει να αξιολογήσει αυτέ τι δυνατότητε που ανοίγονται. Αλλιώ δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Η Κομισιόν θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πλέγμα το οποίο θα εξασφαλίσει την αντιμετώπιση του ρατσισμού κατά το Ρωμά σε όλα τα επίπεδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ρατσιστές κατά το Ρώμα δεν πρέπει να μπαίνουν, δεν πρέπει να μπαίνουν στο κοινοβούλιο μας. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε λοιπόν ότι η μέρα ανάμνησης των Ρωμά θα θεσπιστεί για τις, για τις 2 Αυγούστου ώστε να είναι η μέρα ενθύμησης του ολοκαυτώματος των Τσιγάνων. Την προηγούμενη εβδομάδα και γιορτάσαμε την εβδομάδα των, για του Ρώμα και την ημέρα για του Ρώμα. Υπήρξε μια ευρύτατη πλειοψηφία από όλες τις πολιτικές ομάδες, υπήρξε συζήτηση των επικεφαλιστών κομμάτων, υπήρξαν εκθέσεις, υπήρξαν σεμινάρια, Στο τέλος όμως το συμπέρασμα είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να συμπεριλάβουμε και να ενσωματώσουμε πλήρως τους Ρώμα στην κοινωνία μας. Θα πρέπει να εργαστούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και να αντιμετωπίσουμε τον ίδιο τον κορμό της κοινωνίας μας. Εκεί πρέπει να ληφθούν λοιπόν τα κατάλληλα μέτρα πλέον. Οι απλοί άνθρωποι στο δρόμο, στο λεωφορείο, αυτή τη στιγμή δεν νιώθουν καμία ντροπή όταν εκφράζουν απόψεις κατά τον Ρώμα. Και εγώ το έχω νιώσει αυτό. Έχω ακούσει να μου το λένε πολλοί άνθρωποι στις συναντήσεις που κάναμε. Έχω δει βίντεο που δείχνουν αυτή τη συμπεριφορά των ανθρώπων κατά τον Ρωμά. Και υπάρχουν και οι περιπτώσεις που Ρώμα έχουν υποχρεωθεί να μένουν σε καταβλισμούς όπου είναι σε ένα γκέτο, χωρίς ηλεκτρισμό, νερό, χωρίς ευκαιρίες για υγειονομική περίθαλψη, χωρίς σχολείο για τα παιδιά τους. Είναι μια καταστροφική κατάσταση λοιπόν για τους Ρώμα. Και αν δεν δράσουμε τώρα θα βρεθούμε σε μια κατάσταση η οποία θα είναι αφόρητη, όπου ο κόσμος γύρω μας θα νιώσει φρίκη για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τους Ρώμα. Μπορούμε να έχουμε μια κοινότητα 10-12 εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν κάτω από το <clears throat> κατόφλι της Ένδειας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε λοιπόν να πάρουν τη σκητάλη οι ακροδεξίες δυνάμεις και να χρησιμοποιήσουν αυτή την κατάσταση προς το συμφέρον τους. Τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό και γι' αυτό βλέπουμε την κατάσταση που έχουμε. Εμείς στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών έχουμε διατυπώσει ένα πρόγραμμα για να υπάρξει μια στεναρή στάση για τα θέματα των Ρωμά. Δεν θέλουμε να παραμείνει το status quo έναντι των Ρωμά. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους ηγέτες των πολιτικών ομάδων που έλαβαν μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Ήταν όλοι παρόντες, εκτός από την ομάδα της ALDE ε, Όλοι πάντως συμφωνούν ότι τα θέματα των Ρωμά θα πρέπει να είναι ψηλά στην ε, πολιτική ατζέντα παρά τις προκλήσεις που έχουμε και σε άλλα επίπεδα. Θέλω προσκαλέσω λοιπόν την Κομισιόν να πάρει στα σοβαρά το θέμα αυτό και να προχωρήσει σε δράση. Δεν είναι πια αποδεκτό το 2016 να συνεχίζεται αυτή η απραξία και η αδράνεια ενέτει το Ρώμα. Πρέπει να δράσουμε τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πόστ. Η κυρία Στιτνάσκα έχει το λόγο. Έχει λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Σλοβακία είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες όπου έχουμε πολύ μεγάλη μειονότητα Ρωμά. Στο γύρω στο 49% μάλιστα του πληθυσμού. Λόγω των διακρίσεων και της στόχες ε, έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ δύσκολες καταστάσεις και λόγω των ε, στερεοτύπων που επικρατούν συχνά. Τα παιδιά των Ρωμά πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία και πολλοί έχουν χάσει κάθε ελπίδα για να βρουν ε, απασχόληση. Δεν έχουν κίνητρα και παρά τα κονδύλια που υπάρχουν η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να ενσωματώσει τους ε, ε, πτυχιούχους Ρωμά. Ε, πιστεύουμε πως οι Ρωμά έχουν να παίξουν ρόλο, μπορούν να ηγηθούν των κοινοτήτων μας και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να είναι πιο εμφανίσει οι συμβολή τους. Γι' αυτό και χαίρομαι που την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε έφτιαξε ένα άγαλμα στον Γιάννη Σιμπούλα φυσικού στην Ελβετία και έναν από τους πρωτοστάτες στην δημιουργία του πρώτου κογκρέσου των Ρωμά. Χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία ε, της, της Διεθνούς Μέρας για τους Ρωμά για να δείξουμε πώς η εκπαίδευση μπορεί να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τα σύνορα ανάμεσα στους Ρωμά και τους μη Ρωμά. Κανένας μας δεν μπορεί να αποφασίσει αν θα γεννηθεί γης ή όχι, αν θα γεννηθεί σε μια πλούσια ή σε μια φτωχή οικογένεια. Και χωρίς να υπάρξουν κατάλληλες ρυθμίσεις ε, δεν θα είναι εύκολο να ξεπεραστούν όλες, όλα αυτά τα προβλήματα. Εάν καθυστερήσουμε ε, θα είναι οι επιπτώσεις πολύ σημαντικές για όλους, αρνητικές και σας ευχαριστώ. Κυρία Μλίνερ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ομάδα μας ε, στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία να μιλήσουμε για την Παγκόσμια ημέρα των Ρωμά. Η καταπολέμηση των διακρίσεων σε όλες τις ε, πτυχές της ζωής των Ρωμά θα πρέπει να μας ε, κάνει όλους ε, να μην ξεχνάμε ότι η καταπολέμηση των διακρίσεων και των προκαταλήψεων είναι μία από τις θεμολιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο μόνο μπορούμε να δημιουργήσουμε ίσες ε, συνθήκες διαβίωσης για όλους. Έχουμε δεσμευθεί σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πράξη όμως βλέπουμε ότι δεν τηρούνται αυτές οι αρχές. Υπάρχει αποκλεισμός, υπάρχουν διακρίσεις, δεν υπάρχει πρόσβαση στην αγορά απασχόληση, στο εκπαιδευτικό σύστημα και ε, στην ε, στέγη. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε πλέον να το ανεχτούμε στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει πιο ενεργό δράση και να παρακολουθήσει εάν οι στρατηγικές που έχουν αποφασιστεί υλοποιούνται και αν έχουν και αυτά αποτελέσματα. Πρέπει να δράσουμε και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τηρούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Έρνστ. Νομίζω ότι αυτή η Παγκόσμια ημέρα Ρωμά σήμερα σε αυτή την ε, σχεδόν άδεια αίθουσα είναι κάτι που πραγματικά νομίζω ότι χάνει την σημασία του. Βλέπουμε ότι εδώ και αιώνες ζουν οι Ρωμά στην Ευρώπη, σε, στις περισσότερες από τις ε, χώρες μας. Δεν τους εννοούμε όμως σαν πολίτες των χωρών μας, δεν έχουν τα ίσια δικαιώματα. Η αριστερή λοιπόν της Ευρώπης πολλές φορές βλέπει ότι αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται σαν εχθροί, σαν άνθρωποι οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν ενσωματώθηκαν. Συμμετείχαν όμως στις κοινωνίες μας, στους πολέμους μας και βλέπουμε ότι η ίδια αντιμετώπιση συνεχίζει και σήμερα. Ο Καναδός ε, συγγραφέας ο οποίος αναφέρθηκε σε προσωπικότητες, σε έναν μουσικό, σε έναν συγγραφέα υπερασπιτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανθρώπους που προέρχονται από την κοινότητα των Ρωμά, οι οποίοι θανατώθηκαν και ήταν θύματα του ναζιστικού ολοκαυτώματος. Πότε λοιπόν θα αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν μία κοινότητα σαν πολίτες οι οποίοι ζητούν απλώς ίσα δικαιώματα. Δεν ζητούν ανεξάρτητο κράτος. Ζητούν απλώς να μπορέσουν να ζήσουν όπως εμείς, να ε, ζήσουν με τις οικογένειές τους. Δεν ζητάνε επιπλέον πλεονεκτήματα. Αξιοπρέπεια ζητούν, ίση μεταχείριση. Αυτό λένε και επαναλαμβάνουν. Ίσες ευκαιρίες, τις ίδιες ευκαιρίες με τα δικά μας παιδιά. Σήμερα λοιπόν είμαστε στην ε, δυσάρεστη κατάσταση να πρέπει να αναγνωρίσουμε για άλλη μια φορά ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ίσα δικαιώματα. Δεν μπορούν να εργαστούν σε όλα τα επαγγέλματα. Τους αντιμετωπίζουμε σαν ανθρώπους ειδική κατηγορίας, μουσικούς με κάποιες δεξιότητες. Δεν μπορούν όμως να αντιμετωπιστούν σαν Ευρωπαίοι πολίτες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Ένα θέμα που μας δείχνει ότι ο ρατσισμός και η ξενοφοβία συνεχίζουν να υπάρχουν και ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε στην Ευρώπη για μια κοινωνία με πραγματική αξιοπρέπεια για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις κοινότητες, πολλές φορές κατακαιρματισμένες, μικρές και ζητούν ακριβώς αυτό το πράγμα να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Δεν χρειάζεται λοιπόν να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Θα πρέπει να πούμε ότι η σημερινή μέρα είναι μια μέρα όπως όλες οι μέρες του χρόνου και όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στο Βερολίνο αλλά και αλλού στην Ευρώπη, στο Κοινοβούλιο της Βουδαπέστης όπου υπάρχουν εκπρόσωποι των τσιγκάνων ή στην Ισπανία με την, μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες Ρωμά στην Ευρώπη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να ενσωματωθούν. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες. Θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα και ότι όλοι έχουν δικαίωμα να ζήσουν αξιοπρέπεια στην Ευρώπη. Κυρία Ράιντ και δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι και Ρώμα όλης της Ευρώπη. Η Διεθνή ημέρα των Ρώμα είναι μια ημέρα ανάμνησης, ανάμνησης των αποτροπέων ενεργειών και της δίωξης που υπέστησαν η Ρώμα για εκατοντάδες χρόνια σε αυτή την Ήπειρο. Αλλά είναι και μια μέρα να σκεφτούμε για τις αδικίες που ακόμα αντιμετωπίζουν η Ρώμα κάθε μέρα στην Ευρώπη. Και στο παρελθόν και στο παρόν θα πρέπει να είναι ότι είναι μεγάλη η ευθύνη μας. Υπήρξε ευθύνη μας γιατί δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε μια πλήρως περιεκτική Ευρωπαϊκή Ένωση και να αντιμετωπίσουμε τον ρατσισμό κατά των τσιγκάνων και να εξασφαλίσουμε ίσα δικαιώματα για όλους. Σήμερα μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Μπορούμε να έχουμε μια πολιτική κατά των διακρίσεων. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία που δίνει είδε ευκαιρίε για τη στέγαση, την απασχόληση, την υγεία και την παιδεία. <clears throat> Φαίνεται ότι τα διαφορετικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να μας βοηθήσουν. Αλλά θα πρέπει να ξεπεράσουμε και μόνο τα διαφορετικά ταμεία, γιατί ο αγώνας κατά της διάκρισης δεν αρχεί μονάχα να γίνει σε επίπεδο διαμόρφωσης πολιτικών. Θα πρέπει να φτάσει στην οτροπία της κοινωνίας μας. Ένα παράδειγμα. Οι 11 εκατομμύρια Ρωμά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Όταν εγώ ανοίγω όμως την εφημερίδα βλέπω πάντα το στερεότυπο για τους Ρωμά κάθε μέρα. Αυτό δεν μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τα προβλήματα της διάκρισης και του ρατσισμού κατά τον Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ έχω αγωνιστεί μαζί με τους ακτιβιστές Ρωμά και πολλές φορές ακούω να υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για αυτόν τον αγώνα. Κάποιοι με ευχαρίστησαν βέβαια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εγώ δεν θέλω να με ευχαριστούν. Εμείς θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για την για τον πλούτο που σημαίνει η κουλτούρα των Ρωμά σε όλη την Ευρώπη, για τον αγώνα των ακτιβιστών Ρωμά σε όλη την Ευρώπη και θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους Ρωμά που έχουν ανοίξει τα σπίτια τους, που έχουν μοιραστεί το φαΐ τους μαζί μου και που με, μου επέτρεψαν να είμαι με, μέρος του αγώνα. Θέλω να τους ευχαριστήσω λοιπόν όλους αυτούς που δεν μπορώ να τους απαριθμίσω όλους για το γεγονός ότι μπόρεσα μαζί σας να αγωνιστώ για την περιεκτική ευρωπαϊκή κοινωνία που είναι ανοιχτή στους Ρωμά. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Κάρβερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από όλε αυτέ ε, ε, τις φωνές που έχω ακούσει, θα θυμάμαι πάντα τη φωνή του πατέρα μου που έλεγε ποτέ μην ξεχνάς από ποιο είσαι και από πού προέρχεσαι, γιατί αυτό είναι που σε χαρακτηρίζει. Ήταν Ήταν ε, Ρωμά Αιγύπτος, ήταν ένας χαρακτηριστικός άνθρωπος αυτής της φυλής. ήταν εξαιρετικά σκληρός και νομίζω πως είμαι ο μόνος Βρετανός ενός βουλευτής ε, ρωμανικής καταγωγής και είμαι περήφανος που μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος αυτής της κοινότητας που ζει στο περιθώριο της Βρετανικής κοινωνίας. Ε, στο Συμβούλιο των ε, Ρωμά, των Γύφτων και των Ταξιδιωτών στο Λονδίνο έγραψα και έστειλα και μία επιστολή εκφράζοντα τι ανησυχίε μου όσον αφορά τι πρόσφατε αλλαγέ στην Βρετανία για την νομική προσωπικότητα ενό ταξιδευτή που δημιουργεί προβλήματα στους Ρωμά που ήδη ε, αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικά προβλήματα λόγω ε, λοιπόν διατάξεων. Επίσης έχω γράψει επιστολές ε, στην Βρετανική Επιτροπή Πολέμου γιατί πολλοί Ρωμά χάσαν τη ζωή τους αλλά και τους συγγενείς τους στη διάρκεια των διώξεων των Ναζί. Ποτέ δεν ήταν πιο επίγουσα η κατάσταση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την Βρετανική ταξιδευτική κοινότητα της κοινότητας. Πρέπει να αναλάβουμε αυτή την πρόκληση να την αντιμετωπίσουμε και να μην προσπαθούμε να τα κρύψουμε κάτω από το χαλί και βέβαια δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι θα γίνει κάτι σημαντικό. Η κυρία Επίτροπα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ συναρπαστική συζήτηση. Θα μπορούσα να συνυπογράψω ε, όλα σας τα λόγια και ε, κατανοώ όλα αυτά που είπατε. Η κυρία Σοράγια Πόστ είπε ότι χρειάζονται να γίνουν πολλά και πρέπει να γίνουν τώρα. Η κατάσταση είναι χειρότερη, ε, ε, είναι γιατί έχουμε κάνει πολλά και κάνουμε πολλά, αλλά δεν λειτουργούν προφανώς, γιατί η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Αντίθετα, επιδεινώνεται. Νομίζω ότι αυξάνεται η μη ανεκτικότητα, ε, η έλλειψη ανεκτικότητας. Μάλιστα η Ρωμά είναι μια από τις ομάδες που δέχονται διαρκείς επιθέσεις ε, που τους κοροϊδεύουν και που επηρεάζονται από αυτή την ατμόσφαιρα που επικρατεί στην κοινωνία μας. Γι' αυτό πρέπει να τα καταφέρουμε καλύτερα. Ε, και Σκέφτομαι πολύ για να δω τι, γιατί δεν μπορούμε να καταφέρουμε καλύτερα αποτελέσματα. Πού είναι η φραγμή, ποια είναι τα, ε, η φραγμή και τα εμπόδια, γιατί δεν μπορούν να ενταχθούν οι Ρωμά καλύτερα. Και εγώ βλέπω τρία βασικά προβλήματα. Το ένα είναι ε, ε, είναι το ότι πρέπει να έχουμε συγκεκριμένους στόχους κοινωνική προστασία, απασχόληση, ε, παιδεία. Να δίνουμε την ευκαιρία δηλαδή στα παιδιά και στις οικογένειες με παιδιά και βλέπουμε στα κράτη-μέλη πως αυτοί οι τομείς έχουν ε, υπόκειται σε διαφορετικά υπουργεία και δεν κατανοούν ότι χρειαζόμαστε κοινή δράση. Αυτό αντιπροσωπεύεται, ε, μάλλον τώρα αντικατοπτρίζεται στι εθνικέ στρατηγικέ και ελπίζω πω κάπω θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε σύντομα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι έχω την αίσθηση πω οι πολιτικέ ε, για του Ρωμά γίνονται χωρί του Ρωμά. Πρέπει να τους προσελκύσουμε περισσότερο, να εμπλακούν περισσότερο, διότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς τους ίδιους τους Ρωμά. Και εδώ βλέπω την ανάγκη να υποστηριχθούν περισσότερο οι ΜΚΟ και ορισμένοι, όπως σας το είπατε κιόλα, ότι δηλαδή οι ΜΚΟ και οι κοινότητες που είναι σε καθημερινή επαφή με τους Ρωμά είναι αυτοί που πρέπει να στηριχθούν γιατί συχνά η χρηματοδότηση διακοπτόταν μετά από μια χρονιά. Ενώ το πρόβλημα αυτό είναι μόνιμο. Διαρκώς αναζητούν χρήματα για να μπορέσουν να στηρίσουν τις δραστηριότητες τους, οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε τις ΜΚΟ, ώστε να, να τις χρηματοδοτήσουμε καλύτερα για να μπορέσουν να είναι βιώσιμα τα projects τους. Και το τρίτο πρόβλημα που εγώ διακρίνω είναι ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με ε, καλύτερο τρόπο. Και πάλι μιλάμε για βραχυπρόθεσμα projects, αλλά ενώ μάλλον χρειάζεται πιο μακροπρόθεσμη δράση για να αλλάξει η κατάσταση, διότι δεν είναι μικρό το έργο που έχουμε μπροστά μας αν θέλουμε να αλλάξουν οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα στην κοινωνία. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί σύντομα. Α συνεργαστούμε λοιπόν όλοι μαζί και α είμαστε αρκετά θεραλέοι για να δεχτούμε πω κάνουμε κάτι που δεν λειτουργεί και θα πρέπει να το καταφέρουμε καλύτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε.